περιγράψουμε τέσσερις πράξεις που εγκρίθηκαν μέσα στο πλαίσιο της τακτικής ε, νομοθετικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού του Κοινοβουλίου και οι τίτλοι αυτών των πράξεων θα συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά αυτής εδώ της Συνόδου. Περνάμε τώρα